Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να καθίσετε κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την κοινή συνεδρίαση των επιτροπών μας. χρειάστηκε να καθυστερήσουμε την ε, ε, έναρξη γιατί ε, δεν είχαμε απαρτία. Τώρα όμως έχουμε απαρτία και για τις δύο επιτροπές και έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστώ εν ονόματι της κυρίας Βαλ είμαστε και τα μέλη καλωσόριζω τα μέλη και των δύο επιτροπών και ε, εδώ πρέπει να αποφασίσουμε το πρόγραμμα της δικαιοσύνης ε, επί του οποίου για το οποίο είναι υπεύθυνοι ο Λουίζι Πελιγκουέρ και ο Φιλίπ Κλές. Θα ήθελα να ξέρω αν κάποιος θέλει κάτι να σχολιάσει για διευκρινήσεις ή μπορούμε να προχωρήσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Δεν βλέπω να υπάρξει αντίρρηση, μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως και ε, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Καταρχήν θα ήθελα να κάνουμε μία δοκιματιστική ψηφοφορία για να δούμε αν λειτουργεί το σύστημα. Οπότε ξεκινά η δοκιμαστική ψηφοφορία ηλεκτρονικά για να δούμε αν όλα λειτουργούν κανονικά. Ο κύριος Βοντού δεν έχει ε, την κάρτα. Μπορείτε να βρείτε μία κάρτα στα γρήγορα σας παρακαλώ. Όχι. Υπάρχει όμως κάποιο γραφείο μέσα στο κτίριο το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει. Πρέπει όμως τώρα να ξεκινήσουμε. Έτσι έχει το πράγμα.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 βλέπουμε 26 σήματα. Όλοι ψήφισαν διότι έχουμε 35 κάρτες. Τώρα όμως βλέπω και όλοι, μάλλον αυξάνεται ο αριθμός, αλλά πάρα πολύ αργά. Ψηφίσατε όλοι, ε, πατήσατε όλοι το κουμπάκι σας. Λείπουν ακόμη δύο ψήφοι. Ε, α, τώρα η κυρία Τάιν δεν δούλευε. Κάποιος ακόμη δεν έχει ψηφίσει. Κάποιος δεν έχει πατήσει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε αιωνίως. Οπότε... Βλέπω ότι έχουμε 38 ψηφοδέλτια, ε, κάρτες ψηφοφορίας, ε, από τις 38-37 ψήφισαν ένα όχι. Οπότε ε, μπορούμε να προχωρήσουμε και έτσι ξεκινάμε καταρχήν με την τροπολογία 8 του εισηγητή διότι συνήθως στην νομική επιτροπή έτσι προχωρούμε και παρακαλώ να έχετε κατανόηση ε, και όταν υπάρχουν απλές τροπολογίες ψηφίζουμε διαχειρός και δεν, μάλλον ψηφίζουμε ποιος είναι υπέρ κατά χωρίς να μετράμε τις επιφυλάξεις ε, και ε, θα είναι πολύ πιο απλό έτσι Όσον αφορά βέβαια την ε, τελική ψηφοφορία μετρούνται όλες οι ψήφοι γιατί πρέπει να καταγραφούν στα πρακτικά. Ελπίζω ότι συμφωνείτε με αυτή τη διαδικασία. Τροπολογία 8. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεν βλέπω οπότε προχωρούμε. Η τροπολογία 77 υπέρ. Κατά. Απεφασίστη. Η τροπολογία 78 υπέρ. Κατά. Αποφασίστηκε. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 80 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 9 υπέρ. Κατά. Απερίφθη. 81 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 10 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 82 υπέρ. Κατά εγκρίθηκε 10 υπέρ κατά απερίφθη 11 υπέρ κατά εγκρίθηκε 12 υπέρ υπέρ κατά ε, εγκρίθηκε 11 Τροπολογία 11 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 13 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 14 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 15 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 12 καταπίπτει. Η 86 υπέρ κατά απερίφθη 16 υπέρ κατά ενεκριθεί πλειοψηφικά 13 ε, υπέρ ε, κατά απερίφθη 7 υπέρ κατά απερίφθη ερχόμαστε στη συμβιβαστική 7 υπέρ κατά εγκρίθηκε Τροπολογία 14 υπέρ κατά απερίφθη. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 9 υπέρ κατά απερίφθη. Ε, εγκρίθηκε με συγχωρείτε. Επόμενη σελίδα 93 93 υπέρ κατά Απερίφθη. η 20 διεκπαιρεώθηκε. Μάλλον όχι. Ε, υπέρ. Πρέπει να ψηφίσουμε την 93 υπέρ. Την απορρίψαμε. Ε, με συγχωρείτε. Τώρα είμαστε στην 120 υπέρ. Κατά κατά 120 Α, με συγχωρείτε επανερχόμαστε, γυρίζουμε πίσω γιατί δεν είναι σωστά παρατεθειμένο στο εγγραφό μου 20 υπέρ κατά ενεκρίθη 94 94 υπέρ κατά ενεκρίθη 95 υπέρ κατά δεν χρειά... καταπίπτει δεν χρειάζεται να ψηφιστεί και έτσι ερχόμαστε στη 15 τώρα των γυναικών όπου πρέπει να ψηφίσουν μόνο αυτές τις τρεις γραμμές ποιος είναι υπέρ κατά ενεκρίθη 21 υπέρ κατά ενεκρίθη συμβιβαστική 10 υπέρ κατά ενεκρίθη 97 υπέρ κατά ενεκρίθη 11 υπέρ κατά ενεκρίθη τροπολογία 98 υπέρ κατά απερίφθη 24 υπέρ κατά ενεκρίθη 95 υπέρ κατά ενεκρίθη 16 υπέρ κατά απερίφθη 17 υπέρ κατά ενεκρίθη 26 υπέρ κατά ενεκρίθη 99 υπέρ κατά απερίφθη 18 υπέρ κατά απερίφθη 27 υπέρ κατά ενεκρίθη 100 ε, ο εισηγητής ζητά χωριστή ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Απερίφθη. 19. Υπέρ, κατά. Απερίφθη. 28. Υπέρ, κατά. Ε, νεκρίθη. Ναι, 101. καταπίπτη 102 υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 20 υπέρ κατά εγκρίθηκε 8 υπέρ κατά εγκρίθηκε συμβιβαστική 12 υπέρ κατά εγκρίθηκε τροπολογία 21 υπέρ κατά απερίφθη 107 υπέρ κατά εγκρίθηκε 30 υπέρ κατά ενεκρίθη 31 υπέρ κατά ενεκρίθη 32 υπέρ κατά ενεκρίθη 108 υπέρ κατά αυτό χρειάζεται ηλεκτρονικό έλεγχο. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 108. Δεκαεννέα υπέρ, 22 κατά, άρα κα, ε, καταπίπτει. 9 υπέρ, κατά εγκρίνεται 22 υπέρ κατά απορρίπτεται 109 υπέρ κατά απορρίπτεται 10 υπέρ κατά εγκρίνεται 110 με μία προφορική τροπολογία υπέρ κατά εγκρίνεται 33 υπέρ κατά εγκρίνεται 111 υπέρ κατά απορρίπτεται 34 υπέρ κατά εγκρίνεται 35 υπέρ κατά εγκρίνεται 112 δεν χρειάζεται να ψηφιστεί 113 υπέρ κατά εγκρίνεται 11 υπέρ κατά εγκρίνεται 36 υπέρ κατά εγκρίνεται 12 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβιβαστική 13 υπέρ κατά εγκρίνεται 114 και μόνο το, το πρώτο τμήμα, το δεύτερο τμήμα έχει αποσυρθεί. Πρώτο τμήμα ψηφίζεται υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην 115 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Υπέρ, για να δούμε ξαναψηφίζουμε, κατά. Ναι, προφανώς ε, απερίφθη. 116 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινάει. Η 22 υπέρ 19 κατά εγκρίνεται. 23 ε, υπέρ κατά απορρίπτεται 117 μόνο το πρώτο τμήμα θα ψηφιστεί υπέρ κατά απερίφθη 118 και εκεί μόνο το πρώτο τμήμα υπέρ κατά απερίφθη 119 υπέρ κατά απορρίπτεται 37 υπέρ κατά εγκρίνεται 38 υπέρ κατά εγκρίνεται 39 υπέρ κατά εγκρίνεται 120 υπέρ κατά απορρίπτεται 40 υπέρ κατά εγκρίνεται 121 υπέρ κατά απορρίπτεται 24 υπέρ κατά εγκρίνεται 41 υπέρ κατά εγκρίνεται 42 υπέρ κατά εγκρίνεται τώρα ερχόμαστε στο, στα εκτιμώντας υπέρ 44 ε, υπέρ κατά εγκρίνεται 43 υπέρ κατά απορρίπτεται 45 υπέρ κατά εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 1 14 υπέρ 27 κατά προφανώς απερίφθη συμβιβαστική 1 υπέρ κατά εγκρίνεται Τροπολογία 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά εγκρίνεται 49 υπέρ κατά εγκρίνεται 53 υπέρ κατά απορρίπτεται 51 υπέρ κατά απορρίπτεται 52 υπέρ κατά εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά. Ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 3. «27 υπέρ 17 24 υπέρ 17 κατά εγκρίθηκε 61 υπέρ κατά ενεκρίθη συμβιβαστική 3 υπέρ κατά εγκρίθηκε 57 υπέρ κατά εγκρίνεται 58 υπέρ κατά απορρίπτεται 4 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά εγκρίνεται 5 υπέρ κατά απορρίπτεται 63 υπέρ κατά με συγχωρείτε χωριστή ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα υπέρ κατά στην 63 εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται 64 υπέρ κατά απορρίπτεται 62 υπέρ κατά εγκρίνεται 66 υπέρ κατά εγκρίνεται 69 υπέρ κατά εγκρίνεται 4 υπέρ κατά εγκρίνεται 5 υπέρ κατά εγκρίνεται 6 υπέρ κατά εγκρίνεται 5 υπέρ κατά εγκρίνεται 6 υπέρ κατά εγκρίνεται και πάλι 6 υπέρ κατά εγκρίνεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά εγκρίνεται 7 υπέρ κατά εγκρίνεται 72 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά εγκρίνεται. 74 υπέρ κατά εγκρίνεται. 75 υπέρ κατά εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά απορρίπτεται ε, Τώρα είμαστε στο ψήφισμα, ε, τροπολογία 1 ε, του προπολογισμού υπέρ κατά εγκρίνεται, 2 υπέρ κατά εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στην τελική ψηφοφορία για το κείμενο στο σύνολό του που θα γίνει ηλεκτρονικά για να υπάρξει καταγραφή. Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σαράντα υπέρ, μία κατά, δύο αποχές. Συγχαίρω τους εισηγητές διότι αποφασίστηκε θέλω να ευχαριστήσω εδώ ιδίως του συναδέλφους της Επιτροπής Πληροφοριών που συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Ολοκληρώνεται η κοινή συνεδρίαση και συνεχίζουμε με τη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Θα συνεχίσουμε στο 1G3 ε, και θα ψηφίσουμε στις 45 συνάδελφοι.